Τώρα συνεχίζουμε τη συζήτηση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και δίνω το λόγο στην κυρία Χιμένας Μπεσερέλ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από τότε που ήρθα εδώ στο Κοινοβούλιο, η περάσπιση των θυμάτων ε, ήταν προτεραιότητά μου και όπου και αν είμαι θα είναι προτεραιότητά μου. Οι γυναίκες στην Ευρώπη, τα θύματα βίας μας ζητούν να μιλήσουμε με μία σαφή φωνή και να ενώσουμε τις προσπάθειές μας ε, για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία για το μέγεθος ενός προβλήματος που δεν απλήττει μόνο την Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Η βία κατά των γυναικών δεν κάνει διακρίσεις σε πλούσιες στοχές. Ε, υπερβαίνει οποιαδήποτε σύνορα, χώρο εργασίας, σχολείο, δουλειά. Δεν μπορούν ε, να ξεφύγουν πολλές φορές από τον τόσο κοντινό τους θήτη, τα θύματα. Ε, πολλές είναι οι γυναίκες ε, που μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες ε, έχουν υποστεί σωματική, ψυχική, σεξουαλική κακοποίηση και θα πρέπει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βαδίσουν προς την πλήρη εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Γι' αυτό χρειάζεται μια κοινή στρατηγική. Ως εισηγήτρια ε, επεξεργάστηκα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας ε, των Θυμάτων και στόχος μας τώρα είναι να έχουμε ε, τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης να θέτουμε σε ισχύ εντάλματα που θα αναγκάζουν τον θήτη να είναι σε κάποια απόσταση από τη γυναίκα. πρέπει να μπει ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Εδώ πρέπει να βάλουμε τη γυναίκα στο επίκεντρο και όχι μόνο σήμερα, ε, όλο το χρόνο, για να έχουμε μια πιο ασφαλή, δίκαιη, αξιοπρεπή Ευρώπη. Βλέπουμε ε, τι έχει συμβεί και το χρωστάμε στις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, ε, στα παιδιά τους, να, τις, να μην ξαναγίνουν αυτά ή τουλάχιστον να τα περιορίσουμε. Δέχεστε, λέει πρόεδρος από τον κύριο Έθριτζ, μια μπλε κάρτα. Φρικτό το θέμα αυτό, αλλά στην ουσία πρόκειται για ένα θέμα έλλειψης ε, ηθικής και τιμής στην κοινωνία. Οποιουσδήποτε βλάπτει μια γυναίκα, ε, συμφωνείτε ότι δεν είναι καν άνθρωπος. Ούτε... Φυσικά και συμφωνώ. Απόλυτα συμφωνώ. Και μου αρέσει που μου κάνετε αυτή την ερώτηση γιατί είναι και ένα πρόβλημα παιδείας, που βέβαια σε 1,5 λεπτό δεν είχα χρόνο να το θέσω αυτό το θέμα. Είναι όμως ένα ζήτημα και πρέπει να ξεκινήσουμε και με τους άντρες, ένα θέμα παιδείας. Ε, οι άντρες είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν πιο πολύ να ευαισθητοποιηθούν κατά αυτού του προβλήματος και ίσως και ε, αν όχι ε, περισσότερο από εμάς τουλάχιστον το ίδιο με εμάς τις γυναίκες. Επόμενη μιλήτρια κυρία Αρένα. Ευρωπαϊκή ημέρα της καταπολέμησης της βίας ε, κατά των γυναικών. Είναι αλήθεια ότι αν ε, κοιτάξουμε προς τα δεξιά μας ή προς τα αριστερά μας, ε, είμαστε τρεις γυναίκες, μία τουλάχιστον εξημών υπήρξε, είναι ή θα γίνει θύμα τέτοιου είδους βίας. Ε, και αν δω στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν βλέπω και πολλούς άνδρες ε, δυστυχώς και όντως ε, είναι γεγονός ότι αν οι γυναίκες είναι θύματα βίας σημαίνει ότι υπάρχουν οι θύτες. Και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα και ευχαριστώ τους άνδρες που είναι σήμερα εδώ είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους θύτες όχι μόνο να τους ευαισθητοποιήσουμε αλλά και να τους συνοδεύσουμε και να τους τιμωρήσουμε μία μέρα, μία γυναίκα στις τρεις είναι φρικτό. Και δυστυχώς μιλάμε κάθε χρόνο για αυτό το θέμα, αλλά ε, τα νούμερα αυξάνονται. Ε, δυστυχώς γιατί αυτές η βία δεν μειώνεται, αλλά ευτυχώς γιατί αυτό επιτρέπει στις γυναίκες να είναι περισσότερες, να μπορέσουν να πάνε να καταγγείλουν αυτό που τους συμβαίνουν, να καταθέσουν μήνυση, να τις υπερασπιστεί ένας δικηγόρος, να μπορέσουν να κερδίσουν την υπόθεσή τους ε, στις δικαιοδοσίες τους. Ε, ή τα στοιχεία είναι, μιλάνε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επιτροπές, συζητήσεις και η δουλειά έχει γίνει απαραίτητη και σήμερα κυρία Επίτροπε πρέπει να ενεργήσουμε πλέον. Ε, ε, το θέμα είναι να πάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτή η σύμβαση τη ε, Κωνσταντινούπολη να μπορέσει να κυρωθεί, να κυρωθεί από την Κομισιόν, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα πρόγραμμα δράση. Γιατί δεν αρκεί να κυρώσει κανεί μια, μια, συνθήκη, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει πολιτισμό, δεν υπάρχει διαφορά που να αιτιολογεί το γεγονό ότι σε ορισμένε χώρε μπορούμε καλύτερα να προστατεύσουμε τι γυναίκε από τι άλλε. Πρέπει να εγγυηθούμε ένα κοινό ευρωπαϊκό ε, επίπεδο που θα ευαισθητοποιεί, που θα καταρτίζει τους φορείς, ε, που θα συνοδεύει τα θύματα και τους θήτες αλλά που θα συνοδεύει, ε, που θα μπορεί να τιμωρήσει τους θήτες επίσης. Θέλουμε πλέον αυτή, το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της βίας να γίνει πραγματικότητα. Κύριε Επίτροπε, ελπίζω πως θα ακούσετε αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστώ. Διστάζω να σας ε, διακόπτω καθώς πρόκειται για τόσο λεπτό και σημαντικό θέμα, αλλά πραγματικά θα ήθελα να σας παρακαλέσω <coughs> να κρατάτε το χρόνο σας. Και κυρία Αρένα, για την επίσημη μας ε, κατάλογο μιλητών, έχω δύο άντρες. Έχετε δίκιο κυρία Αρένα για αυτό το θέμα. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ζινάσκα για 1,5 λεπτό. Σα ευχαριστώ. Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Ξέρουμε το μέγεθος του προβλήματος, έχουμε στατιστικά στοιχεία, αλλά σήμερα θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένα νούμερα, όχι ανώνυμα νούμερα. 14% μόλι των θυμάτων της οικιακή βία έχουν το θάρρο να πάνε στην αστυνομία και να ζητήσουν προστασία. Αυτό λέει πολλά για την αξιοπιστία τη αστυνομία στη Σουηδία. 47 Βιασμοί ε, καταγράφηκαν ένα χίλια άτομα, ενώ στην Ελλάδα μόνο δύο, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο διαφορά νοοτροπίας, είναι και διαφορά εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Εάν στραφώ στην αστυνομία θα προστατευθώ, θα βρω μια ομάδα η οποία θα ανεβέσεται και θα ασχοληθεί με το πρόβλημά μου, το πρόβλημα του θύματος δεν θα με αμφισβητήσουν ε, αν λέω αλήθεια ή όχι. Θα, θα καταλάβουν ποιο είναι το πρόβλημά μου και θα με βοηθήσουν να προστατευθώ. Οι δικαστές θα ε, ε, ασχοληθούν και θα προστατεύσουν το θύμα. Το θέμα της βίας κατά των γυναικών δεν είναι μόνο πρόβλημα των γυναικών και των οικογενειών τους, αλλά όλων, πρόβλημα όλων. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν, μην κρίνοντας, απλώς παρακαλώ να μην ρωτάτε τι φορούσε το θύμα ή αν βρισκόταν σε κάποια κατάλληλη γειτονιά. Απλά να ρωτήσετε πώς μπορείτε να τη βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Μπεσέρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επιτρόπε Γιούροβα. Πραγματικά μας ε, συγκλονίζει να το να ξέρουμε ότι μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο, ναι και στην Ευρώπη, κάποια στιγμή στη ζωή τους θα υποστούν σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική βία, κάποια στιγμή στη ζωή τους επειδή είναι γυναίκες και μόνο. Αυτά τα στοιχεία, τα αποτροπιαστικά όμως ε, είναι μόνο ένα κομμάτι, γιατί ε, το 1 τρίτο μόνο των γυναικών καταγγέλει αυτά τα φαινόμενα. Τι κάνουμε όμω, εγώ θα έλεγα να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ριζικά διαφορετικό που θα είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή να επικαιρώσουμε την σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη που είναι το πρώτο ολοκληρωμένο και νομικά δεσμευτικό εγγραφό ε, που λέει ότι η βία κατά των γυναικών και ενδοκαιογενειακή βία είναι σοβαρή επίθεση κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ε, με την σύμβαση αυτή θα μπορούμε να ενδειχνεύουμε, να προλαμβάνουμε και να αποτρέψουμε τελικά τη βία κατά των γυναικών. Διότι έχουμε διάφορε μορφέ. Έχουμε την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, εξαναγκαστικού γάμου, ακροτηρισμό γεννητικών οργάνων, ε, σωματεμπορία κτλ. Θα πρέπει ε, αυτό το εργαλείο ε, που θα βοηθήσει να προστατεύσουμε τα θύματα και να υιοθετήσουμε νομοθετικά και νομοθετικά μέτρα και ποινές να το εφαρμόσουμε. Μέχρι στιγμής 8 μόνο κράτη-μέλη το έχουν επικυρώσει. Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία και Μάλτα 14 το έχουν υπογράψει και είναι στη φάση της επικύρωσης. Είναι μέρα όμως πρέπει να ρωτήσουμε. Βουλγαρία, Εστονία, Ιρλανδία, Τσεχία, Κύπρα, Κύπρο και λοιπόν. Γιατί ούτε καν έχουν υπογράψει αυτό το, αυτή την σύμβαση. Είναι μια Ωραία μέρα σήμερα το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Κομισιό να δεχτεί αυτή την εντολή και η νέα Λετωνική Προεδρία ε, να πάρει τα ενία από τον Ιανουάριο. Ε, είναι ένα σημείο αναφοράς ε, για την πρόσπιση της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να έχει μία φωνή κατά ε, της ε, τιμωρία των γυναικών αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να διώκεται και πρέπει να στηριχθούν όλοι όσοι βοηθούν τις γυναίκες, όπως ο δόκτωρ Μουκάμπε. Θα πρέπει να κατηγορήσουμε, να, να καταγγείλουμε την ανισότητα αυτό που συνεχίζει να μας προκαλεί ντροπή. Um, Σε ευχαριστώ. Έχουμε, έχουμε μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρες. Η τραγωδία που συζητάμε σήμερα εδώ έχει επίσης ε, πολιτιστική προέλευση προέρχεται από ένα, μια κουλτούρα που θεωρεί υποδέστερη τη γυναίκα. Σήμερα όμως είχαμε τον αρχηγό της Εκκλησίας που εμποδίζει, απαγορεύει την ιεροσύνη στις γυναίκες και μάλιστα εξακολουθεί να ισχύει στο Ευαγγέλιο αυτή η παράγραφος όπου η γυναίκα εορκίζεται υποταγή στον άνδρα. Ε, αυτό επιτείνει αυτό που λέμε, δηλαδή τη βία κατά των γυναικών. 30 ε, δευτερόλεπτα έχετε για την ερώτηση, συνάδελφε. Έχετε και εσείς τώρα 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Σήμερα ο Πάπας μας μίλησε για αξιοπρέπεια και νομίζω ότι αυτή η αξιοπρέπεια ε, είναι πάνω απ' όλα. Το να μιλάμε για την αξιοπρέπεια ε, των ανθρώπων σίγουρα έχει να κάνει με τους περισσότερους, με τον μεγαλύτερο πληθυσμό που είναι γυναίκες. Και το είπε ξεκάθαρα ο Πάπας, δεν υπάρχει τίποτα πάνω από την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, των προσώπων συγκεκριμένα. Μπιόρκ για 1,5 λεπτό. Μάρα Μπιόρκ. Ε, for the day being. Ε, jag skulle vilja börja med att tacka alla de kvinnor som har jobbat outtröttligt före oss. Ε, είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να μένει μόνιμα στην ημερήσια διάταξη. Οι προηγούμενοι ομιλητές ε, και κυρίως η Εύα Βένσο που είναι στην Επιτροπή Γυναικών ε, θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί η δουλειά της Επιτροπής Γυναικών είναι αυτή που μας βοηθάει και μας βοηθά να προχωρήσουμε. Είναι προφρικτέ αυτές οι στατιστικές, ε, Φρικτά τα νούμερα δείχνουν μια παράδεκτη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα όπου οι γυναίκες δέρνονται γιατί επειδή απλά είναι γυναίκε, γυναίκε και κορίτσια τα οποία δεν έχουν ε, κανένα δικαίωμα γιατί οι τα δικαστήρια δεν καταδικάζουν τους δήμιους τους. Ε, πώς μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να μην συνεχίζεται. Είναι ένα θέμα ισχύω ε, και εξουσίας που εισάγει ανισότητα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες και εκεί θα πρέπει να παρέμβουμε. Ο πολιτισμός ε, όπου το σώμα της γυναίκας δεν της ανήκει, ε, ε, μια κουλτούρα όπου γίνονται διαρκώς εξιστικά σχόλια έναντι γυναικών και κοριτσιών. Όλοι γνωρίζουμε κάποια γυναίκα που έχει βιαστεί και γνωρίζουμε όλοι και κάποιον βιαστή. Όταν τίθεται το θέμα προσυζήτηση δημοσία, θα πρέπει πια να δράσουμε, να ενεργήσουμε, να ακούσουμε κόσμο που να λέει ναι, πρέπει να δράσουμε σε νομοθετικό επίπεδο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και όλα τα κράτη-μέλη να την κυρώσουν επίσης. Πρέπει να πάψει πια αυτή η βία. Ευχαριστώ κυρία Μπιόρκ. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ουρτασούν. Κυρία Επίτροπε, ίσως δεν το λέμε συχνά, εγώ θέλω να το πω όμως, η ανισότητα και η άνηση κοινωνία στην οποία ζούμε φυσικά και είναι μοχλός για την αύξηση της βίας ε, και οι περικοπές των δημοσίων υπηρεσιών είναι ένα πρόβλημα που ακριβώς ε, ε, οξύνει το φαινόμενο της βίας. Δεν θέλω να επαναλάβω τα στοιχεία που έδωσαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά 25 Νοεμβρίου σήμερα και γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε ένα ειδικό ε, νομικό μέσο για την καταπολέμηση της βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπατε ότι έχουμε τη στρατηγική περισσότερα των φύλων και άλλα εργαλεία. Όχι όμως ένα συγκεκριμένο θετικό εργαλείο ακριβώς για αυτό το θέμα και ελπίζω κάποια στιγμή να το έχουμε. Θέλω να πω επίση ότι αυτό που είπατε δεν μου άρεσε για το παρατηρητήριο. Είπατε δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Εγώ λέω ότι είναι. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μάστιγα. Και σε ό,τι αφορά τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, συμφωνώ ότι πρέπει να εγκριθεί από όλα τα κράτη-μέλη και να επικυρωθεί. Πρέπει να πω ότι αυτή η σύμβαση και η επικύρωσή του δεν υποκαθιστά το γεγονό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε ένα ειδικό νομοθετικό μέσο. Γι' αυτό θέλω να σα συγχαρώ και να σα συστήσω από τη δική σα θέση τώρα να προωθήσετε τη δημιουργία αυτού του μέσου το οποίο τόσο είναι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, Αγιούτο. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας έναντι των γυναικών. Εδώ είμαστε προσπαθώντας να πείσουμε την Επιτροπή να νομοθετήσει για αυτό το θέμα. Αν και ορισμένες αρμοδιότητες ε, βαραίνουν τα κράτη-μέλη, εμείς θα περιμέναμε μια πρωτοβουλία να ξεκινήσει από την Κομισιόν τουλάχιστον για τα όσα αφορούν τις δικές της αρμοδιότητες. Αν θεωρήσουμε ότι άριθμα κράτη μεταξύ, μεταξύ αυτών και Ιταλία έχουν ήδη κυρώσει τη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης και έχουν νομοθετήσει σχετικά. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι μόνο σωματική. Πολύ συχνά είναι και κυρίως είναι ψυχολογική και συνήθως εντός των ε, ε, οικιακών τυχών και ε, παρασύρει και τα ανήλικα του σπιτιού. Υπάρχουν διάφοροι κόδωνες κινδύνου που συνήθως όμως δεν εισακούγονται γιατί η νομοθεσία είναι ελλειπής. Αν είχε υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τραγωδίες. Σκέφτομαι την υπόθεση, την περίπτωση της Λουτσία Μίγκολη που ο πρώην αραβωνιαστικός της ε, την ε, ε, περιέλωσε με οξύ. Άλλος που, που σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των παιδιών του που ήταν μόλις 5 και 6 ετών. Μην ξεχνάμε πως τέτοιου είδους δολοφονίες είναι σε αύξηση. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε ότι στην έκθεση Εύρες μόνο στην Ιταλία υπήρξαν 179 τέτοια περιστατικά. 2013. Έχετε ξεπεράσει τον χρόνο σας, δεν μπορώ να σας αφήσω περισσότερο. Σας έχω προειδοποιήσει. Είναι πολλοί εκείνοι που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία Καριστιά και προσπαθώ να αφήσω το δυνατόν περισσότερους αδέρφους να συμμετάσχουν στη συζήτηση. κυρία Μορβάη έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Άνθρωποι που φοράνε καλά και ακριβά κοστούμια, ακριβά ρολόγια, περπατάνε στους δρόμους το βράδυ και κινδυνεύουν βέβαια με τα ακριβά τους ρούχα να προσελκύσουν τους κλέφτες. Αυτό θα μας έλεγε η Επιτροπή. Αυτό θα λέγαμε ότι αν δίνεται κανείς με ακριβά ρούχα κινδυνεύει από βία. Και όμως αυτό έχει κάνει σε αντίστοιχο βίντεο η Επιτροπή για τη βία σφαίρα των γυναικών στη χώρα μου. Εγώ θα συνιστούσα έναν διαφορετικό καλύτερο φίλμ. γιατί υπήρξαν εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχών που έλεγαν Μάλλον θα θέλαμε να δούμε εκπροσώπους των αστυνομικών αρχών να λένε ότι όποιος έχει διαπράξει κλιμαβία στις φάρος γυναίκας θα πρέπει να συλλαμβάνεται να προσάγει τη δικαιοσύνη και να καταδικάζεται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να διαπιστώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό δεν θεωρεί ε, ε, όριμο την ε, στιγμή για να προτείνει νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με εντυπωσιάζει σήμερα, με κάνει να απορώ. Θα ήθελα να θυμίσω στην Κομισιόν ότι η ίδια έχει αναγνωρίσει στη βία κατά των γυναικών το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη μιας πραγματικής ισότητας των φύλων πώς θα συμβάλλουν, πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε την συμβολή, την έλλειψη της συμβολής της κυρίας Βαρβανόβα, στις δυσκολίες των κρατών μελών, θα τα ρίξουμε όλα. Ε, πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι όλοι, το Κοινοβούλιο επιμένει εδώ και καιρό ώστε να υποβληθεί επιτέλους μια οδηγία, μια πρόταση οδηγίας που θα θέτει τέλος στην ατιμορρησία της γυναικοκτονίας που θα ευνοεί το κράτος που θα στηρίξει ε, τα θύματα και που θα βελτιώσει την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη. Επίτροπε, εσείς ε, στην αρχή της ε, παρέμβασής σας ε, αναφέρατε διάφορα στοιχεία. 33% των γυναικών είναι θύματα ήδη από τα 15 τους χρόνια και 20 με 25% των γυναικών έχουν γίνει θύματα ψυχολογικής ή σωματικής βίας τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Όμως όλα αυτά τα στοιχεία δεν αρκούν για να προστατευτούν τα θύματα. Δεν νομίζετε. Εγώ είμαι πεπισμένη πως αυτό το νούμερο είναι επαρκή για να αιτιολογηθεί η εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού μέτρου νομοθετήματος που θα θεσπίζει κοινέ αναφορές. Σήμερα, αυτή τη σημαντική μέρα, θα πρέπει να πούμε αλήθεια αν υπάρχει βία ή όχι και να ενεργήσουμε για να καταπολεμηθεί. Είναι θέμα πολιτισμού και δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι παρακαλώ να είσαστε όλοι προσεκτικοί με το χρόνο και να τον σέβεστε. Η κυρία Μπλίνκεβιτσούτα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, πατρίδα μου τη Λιθουανία έπεσε θύμα βιασμού και βίαιου φόνου μια κοπέλα, φοιτήτρια, 20 ετών. Ένα κορίτσι άκακο, όπως μας είπε και η μητέρα της. Αυτό συμβαίνει στη μία σε τρεις γυναίκες στην ανεπτυγμένη και προοδευτική μας Ευρώπη. Μία στις τρεις πέφτουν θύματα ε, βιασμού στη διάρκεια της ζωής τους. Μία στις 17 φωνεύεται κάθε μέρα είναι δυνατόν εμείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λησμονήσουμε το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό επιμένουμε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της βίας της των γυναικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί κάθε κράτος χωριστά να καταπολεμήσει τη βία γιατί χρειάζεται ο συντονισμός σε όλους τους τομείς, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δικαιοσύνη, την παρακολούθηση, την υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους τομείς και χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της βίας βάρο βάρος των γυναικών. Μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε με φυστάμενες δομές και όχι θεσπίζοντας νέες δομές. Μπορούμε να επεκτείνουμε δηλαδή τη δράση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Ευχαριστώ πολύ και τώρα παρακαλώ να λάβει το λόγο η κυρία Βυσνιεύσικα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μας επισκέφθηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώτος, και μας είπε ότι αν με το Θεό πέφτουμε, περιπέφτουμε στη βία. Ξεχνάμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η βία στρέφεται κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πέφτουν κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο οι γυναίκες θύματα της βίας αυτής βία εκδηλώνεται και στα ανεπτυγμένα λεγόμενα κράτη. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με βία εις βάρος και των γυναικών στο Ισλάμ αλλά και στην Ευρώπη. Πρέπει να λάβουμε μέτρα, αλλά τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να είναι απλά νομοθετήματα. Δεν λύνουν τα προβλήματα οι οδηγίε. Υπάρχουν αρκετέ ρυθμίσει, ανάλογα με τις παραδόσεις και τα έθιμα σε κάθε κράτος. Δεν υπάρχει λόγος σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εισαχθούν νέε οδηγίε. Τα κράτη-μέλη πρέπει απλώ να υλοποιήσουν τις εφιστάμενες, την εφιστάμενη νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ, Μπίρτερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εκδόθηκε φέτο μια έκθεση τη Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μα δείχνει ότι η έκταση των, ε, των βιοπραγιών ε, εις βάρος των γυναικών είναι τέτοια που και οι αρχές ακόμη καταστολής, οι αρχές της τάξης γίνονται πλέον ε, πολύ πιο χαλαρές έναντι τέτοιου φαινομένου. Είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξουαλικής βίας ε, από ε, εταίρο σύντροφο ή μέλος της οικογένειας. Χρειάζεται λοιπόν μια νομοθετική πρόταση μέχρι το τέλος του 2014. Ευρωπαϊκή δράση, ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο έτσι μας λέει η υπηρεσία. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει στα τέλη του Νοεμβρίου σχεδόν και δεν έχει γίνει τίποτα. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωράει σε μέτρα για την καταπολέμηση του ακροτηριασμού, του σεξουαλικού ακροτηριασμού των κοριτσιών. Πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, γιατί βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να αναπτύσσεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γυναίκες και κορίτσια Ευρωπαίες πέφτουν θύματα αυτού του ακροτηριασμού ή τη βία ή τη εκμετάλλευση ή του εμπορίου εις γυναικών. Πρέπει αυτό το φαινόμενο να καταπολεμηθεί με αποφασιστικότητα από όλους μας. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μεμονωμένα, αλλά ως κομμάτι ενός ευρύτερου προβλήματα ή την στάση τη της κοινωνίας έναντι των γυναικών. Και χρειάζεται δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο κρατών μελών. Χρειάζεται δράση τώρα. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα λάβει το λόγο η κυρία Κούνεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα με επιτρέψετε να κρατήσω στη θέση μου να μην σηκώνω με όρτια λόγω την κατάστασή μου. Τα στοιχεία της σωματική και ψυχοϊκή βία είναι συντριπτικά. Περίπου 13 εκατομμύρια γυναίκες δηλώνουν θύματα σωματικής βίας, δηλαδή το 7% των Ευρωπαίων γυναίκων ηλικία 18 έως 74 ετών. Η βία κατά των γυναικών έχει πολλά πρόσωπα, δεν γνωρίζει σύνορα και τάξεις, επιβάλλεται με σκληρούς άντρες αντισόπιτους τρόπους. Έχει βιωθεί μέσα στην οικογένεια, στην κοινωνία και τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά στην εργασία. Προσωπικά βίωσα σκληρή βία για να σταματήσει η εκδίκηση των δικαιωμάτων μια τάξη ανθρώπων για να μην ακουστεί η φωνή του. Όμω τώρα αναβιώνει και ένα νέο κίνημα οικονομικής βίας στην Ελλάδα η εργοδότη ζήτησε από εργαζόμενοι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη να διακόψει την κοίηση ή αν θέλει να έχει δουλειά. Φαινόμενα όπως αυτά εργαζομένων γυναικών που φοβούνται να δηλώσουν την εγκυμοσύνη τους γιατί ο εργοδότης δεν επιθυμεί να δεσμευτεί πως δεν θα τις απολύσει για τους 18 μήνες που ακολουθούν μετά το τουκετό είναι η καθημερινότητα στις χώρες που επιβλήθηκαν τα αυστηρά δημοσιονομικά προγράμματα. Να αντιμετωπίσουμε τη βία που στρέφεται τόσο απρόκλητα ακόμη και ανάντια στη μετρότητα με μια νομοθετική ρύθμιση με συνδυασμό με την κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη γνωστή σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο νομικής προστασίας. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Επόμενο κυρία Ντέλη. Ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, 62 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους. Είναι σκανδαλωδώς υψηλά τα νούμερα αυτά. Δεν μπορούμε να τα γνωρούμε πλέον. Και εσείς κυρία Επίτροπε δεν μπορείτε απλώς να μας λέτε ότι το ανακαλύψατε. Ποια είναι λοιπόν τα ζητήματα, πώς είναι δυνατόν ο βιασμός να μην αναγνωρίζεται ακόμη ως ποινικό αδίκημα σε κάθε κράτος μέλος. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι το 2014 η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης που εξασφαλίζει ένα πλήρες πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων, για την προστασία από τον ε, Δήμιο, για την αποτροπή των εγκλημάτων να μην έχει κυρωθεί παρά μόνο από 8 κράτη-μέλη. Πώς είναι δυνατόν εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς ως να μην έχετε κάνει μια πρόταση για νομοθέτημα ζήτημα. Χρειάζεται ένα παρατηρητήριο τη βία τη βάρα των γυναικών, ένα πλαίσιο δεσμευτικό, νομικό δεσμευτικό πλαίσιο, ώστε άνωθεν να επιβληθούν τα μέτρα πρόληψη και πρέπει να ασκήσετε πίεση εσεί τα κράτη-μέλη για να ακυρώσουν τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη και κατά λίγο δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει πλέον να βγουν οι γυναίκε από τη ζώνη αυτή χωρί δικαιώματα στην οποία του έχει περικλείσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πάρκερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα που δεν θα αναφέρει κανείς σας είναι η πλήρης ελευθερία διακίνησης εντός Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή έχουμε την ανοιχτή πόρτα αυτή την πολιτική στη μετανάστευση, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ποινικό ή εγκληματικό επάβαθρο των εισερχόμενων που έχουν παρελθόν λοιπόν καταχρήσεων, κακοποιήσεων, βία ή να είναι μέλη εγκληματικών σημεριών, να έχουν κακοποιήσει γυναίκε. Όλοι αυτοί οι εγκληματίε μπορούν να μπουν χωρί ε, να του ρωτήσει κανεί ε, τίποτα ε, πολύ ελεύθερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Χάρη στου ωραίου κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τρέλα φυσικά όλα αυτά. Πριν αρχίσετε λοιπόν να ζητείτε ακόμα πιο άχρηστη γραφειοκρατία Καλύτερα να πάψουμε στους εγκληματίες ε, και σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί να τους παρέχουμε την ελευθερία πρόσβαση στις χώρες μας. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι πραγματικός έλεγχος στα σύνορα. Με τους ελέγχους αυτούς να δυσκολεύουν μέλη εγκληματικών συμμοριών, διακινητές προσώπων ή με ιστορικό βίας να μπουν στις χώρες μας. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Μάγερ για ένα λεπτό. Ή μάλλον υπάρχει μπλε κάρτα. Ζητώ συγγνώμη, θα τη δεχτείτε. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κυρία Ρενά, όταν ακούω αυτά ε, που ακούω βγαίνω από τα ρούχα μου, πραγματικά. Ε, ξεκινάμε ε, και συνδέουμε τους βιασμούς με την είσοδο μεταναστών. Είναι απαράδεκτο να βγαίνει από το σώμα μιας γυναίκας αυτό. It was more a statement. Πιο πολύ περιδηλώσει επρόκειτο. Τέλο πάντων, θα δώσω το λόγο να απαντήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Απλά σα ευχαριστώ την προσοχή. Σε ένα τραγικό φόνο πριν από δύο μήνε, μια νεαρές γυναίκα στη χώρα μου, η οποία έχασε τη ζωή τη, ε, καταδικάστηκε, νομίζω, ένα Λιθουανό ήταν αυτό, που είχε ήδη καταδικαστεί για φόνο. Αλλά αυτό ο άνθρωπο είχε μπει ελεύθερα στη χώρα μα. Ίσως έτσι θα είχε σωθεί μια ζωή. Ε, επαναλαμβάνω, ίσως θα έχει σωθεί μια ζωή, ίσως θα έχει σωθεί μια ζωή. Εάν υπήρχαν τα θεσμικά αντίβαρα. Δεν πρέπει τον έλεγχο των συνόρων ε, και την περιορισμό των εγκληματιών να το υποτιμούμε ως μέτρο. Πρόεδρος, θα δώσω δυνατότητα ε, σε ένα δεύτερο σάλιφο να θέσει ερώτημα στο πλαίσιο της μπλε κάρτας. Παρακαλώ. Λέτε ότι μπορείτε να σταματήσετε την ελεύθερη κυκλοφορία. Πώς θα πείτε ας πούμε σε έναν Σκοτσέζο, μάλλον πώς θα απαγορέψετε έναν Σκοτσέζο εγκληματία να πάει στο Λονδίνο ή έναν ε, από το Λονδίνο να πάει στη Βόρεια Ιρλανδία. Απάντηση. Δεν είναι θέμα να ελέγχουμε αυτό. Αλλά να ξέρουμε αυτοί που έχουν ποινικό μητρό, που βρίσκονται και τα θύματα, τα αθώα, να τα προστατεύσουμε. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ζωτικό να προστατεύσουμε τα θύματα. Όχι, δεν το δέχομαι. for that exchange. We move to our next Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Επόμενο ο μιλητή Μάιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, μπορεί κανείς να αισθάνεται συγκλονισμένο σε αυτά τα γεγονότα. Η ισότητα ανδρών και γυναικών δεν είναι κάτι το φυσιολογικό. Και δεν δικά μου λόγια, είναι λόγια του Τούρκου Προέδρου, κ. Ερντοάν, τις τελευταίες ημέρες. Μας είπε λοιπόν ότι δεν είναι φυσιολογικό πράγμα ισότητα ανδρών και γυναικών. Εδώ λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε και δυστυχώς στον 21ο αιώνα υπάρχουν ακόμη τραγικές περιστάσεις ή υποθέσεις βίασης βάρος των γυναικών. Όχι μόνο βέβαια στην Τουρκία όπου 34% των γυναικών έχουν πέσει μια φορά στη ζωή του τουλάχιστον θύμα ε, βίας. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στη Σουηδία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία. Ρότενχαμ, παραδείγματι. Χιλιάδε κορίτσια είχαν πέσει θύματα βία για δεκαετίε στο Ρότενχαμ. Ξέρετε σε τι οφείλεται όλο αυτό. Στο ότι πρέπει καταρχάς να βγάλουμε τα γυαλιά του πολιτικού ορθού και να μιλήσουμε ξεκάθαρα για την μετανάστευση ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια τελείως διαφορετική ιδέα και αίσθηση για το τι σημαίνει γυναίκα. Ευχαριστώ πολύ για 1,5 λεπτά, αισθαράς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσο και αν προσπαθούν αυτοί να το ε, σκοτώσουν αυτό που έχουμε μέσα μας, δεν θα το καταφέρουν. Ε, όσο μπορώ θα αντιστέκομαι, θα βρω τη δύναμη μέσα μου. Η Ενίσα τα είπε αυτά ε, είναι μία από τους επιζήσαντες, επιδόσαντες από τον πόλεμο στην Βοσνία. Σίγουρα η βία μπορεί να έχει πολλές μορφές, οικονομική, σωματική, σεξουαλική, σωματεμπορία, ε, εξαναγκασμός σε γάμο. Και είπαμε ότι μία στι τρεις νίκες ε, δέχονται ότι έχουν πέσει θύμα βίας κάποια στιγμή στη ζωή τους. Αλλά μιλάμε και ε, για συμπεριφορές και των εφήβων. Έχουμε την νέα τεχνολογία οι έφηβοι e πολλές φορές είναι θυσμένοι ε, στις νέες τεχνολογίες ε, στο διαδίκτυο, αλλά δεν καταλαβαίνουν ε, πολλές φορές ότι μπορούν να πέσουν θύμα και βίας και μέσω του, του κυβερνοχώρου. Υπάρχουν 2,6 εκατομμύρια τέτοια κρούσματα βίας κατά των γυναικών γενικώ και παρόλα αυτά δεν έχουν μια στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θέλουμε να εναρμονίσουμε τα συστήματα των 28 κρατών μελών. Και η σύμβαση αυτή ε, της είναι, είναι πολύ σημαντική. Πρέπει όλη η κοινωνία να ε, ευαισθητοποιηθεί. Θέλουμε πολιτικές, εταιρική σχέση, να σπάσουμε τη σιωπή, να διώξουμε τους ε, θύτες ε, και βέβαια ε, τα ευάλωτα άτομα, τα παιδιά, τα κορίτσια, τους ομοφιλόφιλους, άτομα με αναπηρίες, πρέπει να τους προσέξουμε. Κύριε Ροντρίγκης τώρα έχει το λόγο. Queria falar da Convenção de Istambul, que consagra, os direitos das mulheres. Πρέπει να ακυρωθεί η σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης που προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχουν όμως κάποιες αμφιβολίες. Ήδη είπαμε στην Ευρώπη 100 ε, ε, εκατομμύρια έχουν γίνει θύματα βίας βρίσκονται σε κίνδυνο αυτή, για αυτή την, την, ε, την, ε, τον ακροτηριασμό των γενετικών ε, οργάνων πολλές γυναίκες, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης οι γυναίκες θα είναι σίγουρα πιο προστατευμένες. Η αλήθεια είναι όμως πως ο αριθμός των θυμάτων της βίας ακόμα ε, δείχνει ότι ακόμα δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Τα νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν από πλευρά των κρατών που κύρωσαν τη συνθήκη τη Κωνσταντινούπολη. Ε, συμπληρωματικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν, ε, πρέπει να γίνουν μηχανισμοί ε, εντοπισμού και θα επιβληθούν ποινές. Ε, η Κομισιόν έχει τη δύναμη να πείσει τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση τα κράτη-μέλη τα ίδια. Θα πρέπει αυτή η σύμβαση ε, όντως να εφαρμοστεί και αν δούμε και τον ίδιο το πρόεδρο της Τουρκίας που θεωρεί ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι ενάντια στην φύση. Ένα λεπτό, Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κανεί εδώ δεν είναι υπέρ τη βία κατά των γυναικών βέβαια. Βεβαίως. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να ενωθούμε και να προτείνουμε τρόπους που πιστεύουμε ότι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε, να κάνουμε κάτι. Τα 28 κράτη-μέλη έχουν συνομοθεσία που καθιστά ποινικό αδίκημα την βία κατά των γυναικών, αλλά δεν την επιβάλλουν πάντοτε. Ας ενωθούμε, έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά α κάνουμε και κάτι παραπάνω. Πριν από 30 χρόνια στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της αστυνομίας της ε, του Λονδίνου είπε ε, «Τα δέσποτα σκυλιά και, και εκεί βία». Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να αντιμετωπίσει η αστυνομία μας. Όμως κατά μέσο όρο ακόμα και σήμερα δύο γυναίκες ε, σκοτώνονται κάθε μήνα από την οικιακή βία. Έχουμε ποινικοποιήσει τους καταναγκαστικούς γάμους, έχουμε περάσει διάφορες νόμους που επιτρέπουν στην αστυνομία να αποκαλύπτουν πληροφορίες σε σχέση με το προηγούμενο ιστορικό βία των, των εταίρων. εταίρων. Οπότε, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, ας ε, ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ας βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε ώστε να πάψει αυτή η κατάσταση και να μην ε, επιτιθέμεθα μόνο εναντίον της επιτροπή. Σας ευχαριστώ και επαναλαμβάνω την απροθυμία μου να διακόψω αυτή τη συζήτηση, αλλά είπα ότι έχουμε πολλούς ομιλητές και έχουμε ήδη καθυστερήσει. Επόμενο ομιλητής, ομιλήτρια για ένα λεπτό είναι η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη Χρειάζεται τη συμμετοχή όλων των εταίρων στην υποστήριξη. Πρέπει να ε, καταπολεμηθεί η βία κατά των ε, γυναικών και των ε, εφήβων, κοριτσιών. Δεν έχουμε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Έχουμε καταφέρει αλλού, παραδείγματος χάρη για άλλους μορφές βίας, αλλά δεν έχουμε καταφέρει εδώ να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα. Αν θέλει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, στατιστικά στοιχεία, κοινέ αξίε, κανένα ευρωπαϊκό κράτο δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το θέμα να το θεωρεί ιδιωτικό ζήτημα. Η έλλειψη ενεργών πολιτικών, η μη συμπερίληψη τη βία κατά ε, των γυναικών ε, στα θέματα που απασχολούν ένα κράτο, ε, ουσιαστικά παραβιάζει τι συνθήκε και γι' αυτό σα ζητώ. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να υποβάλλετε κυρώσει στι κυβερνήσει που το πράττουν αυτό. Και επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Κοσλόφσκα για ένα λεπτό. Ενάμιση. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Η βία είναι έγκλημα και αφορά όλο τον κόσμο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με αποτελέσματα μακροχρόνιας βίας εις βάρος των γυναικών και διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Πρέπει πια να αλλάξουμε λοιπόν και νοοτροπία. Συμφωνώ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη βία, για την αντιμετώπιση της βίας βάρος των γυναικών, γιατί και αυτή μιλάει και για ισότητα μεταξύ των φύλων και για τη μετώπιση των προβλημάτων. Κυρίε και κύριοι, οι προσπάθειες μα στα κράτη-μέλη χρειάζονται και παρακολούθηση. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε συγκρίσιμα δεδομένα που να μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Χρειαζόμαστε ε, μια κοινή μέθοδο συλλογής και ανάγνωση των δεδομένων και γι' αυτό θέλω να απευθύνω έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα φέρει μια, να εκδοθεί μια σύσταση ή αργότερα και μια ε, οδηγία η οποία θα μπορούσε να αναρμονίσει τη μέθοδο αξιολόγηση, συλλογή στοιχείων που έχουν να κάνουν με τη βία των γυναικών. Ιδάλλως, ναι, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιώτοβα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η σιωπηλή κραυγή τη Βία. Έτσι ονομάστηκε ένα φόρουμ στην Βουλγαρία, ένα φόρουμ που στόχο έχει να καταπολεμήσει τη διέσβαρση των γυναικών. Και έχουμε να κάνουμε με ένα τίτλο που δεν αποτελεί απλώς μια θλιβερή διαπίστωση. Έχουμε να κάνουμε με έναν τίτλο ο οποίο εκδηλώνει ταυτόχρονα και τη βούλησή μα να καταπολεμήσουμε αποφασιστικά το πρόβλημα αυτό. Και γι' αυτό στρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επίτροπο. Δεν χρειαζόμαστε νέα όργανα, νέε υπηρεσίε. Χρειαζόμαστε ε, νομοθεσία η οποία θα μπορεί όχι να προβλέπει ποιο θα είναι το θύμα, αλλά να προλαβαίνει τα εγκλήματα. Δεν έχουμε αρκετά μέσα. Είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αρκούν τα μέσα που έχουμε στη θέση μας. Και πρέπει να προχωρήσουμε σε ταχύτατη κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολη. Και αυτά τα οποία περιλαμβάνει θα πρέπει να μεταφραστούν σε πράξεις. Έστω και αν ο κύριος Ερντοάν ο ίδιος ε, που φιλοξένησε τότε εκείνη τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης λέει πως ο θέση τη γυναίκας είναι στο σπίτι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια νέα οδηγία, μια νέα νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ για μισή λεπτό. Η κυρία Κομοντίνη. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, 30 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας ε, και πολλά εκατομμύρια γυναικών είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας ε, στην περίοδο που προηγήθηκε τις, ε, στο 12 μήνε προηγήθηκαν τις έκθεσεις της αρμόδιας υπηρεσία. Εδώ η βία των γυναικών είναι σημάδι στο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ουλή και αφορά όχι, όλα τα, όχι ένα κράτος μέλος, αλλά όλα τα κράτη-μέλη. Μόνο από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εάν ενώσουμε τις φωνές μας, αν ενώσουμε τη φωνή τις δράσεις μας. Η βία σφαίρος των γυναικών είναι διαδεδομένη και εκτεταμένη. Έχει να κάνει βέβαια με παραβάσει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια ένωση λοιπόν στηριγμένη στην ε, προστασία και το σεβασμό τη ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα εγκλήματα αυτά μεμονωμένα. Πρέπει να συμμετάσχουν οι πάντες, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορέ, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, φορείς, εθνικές αρχές και όποιος άλλο. Χρειάζεται μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο υγειονομικής περιθάλψης, συνοχή, υποστήριξη. Και πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε υφιστάμενο μέσο ώστε να εξασφαλίσουμε μέτρα προστασία και ταυτόχρονα να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άντρε κοιτάνε τι γυναίκες τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ένα τον άλλον. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπορζάν. Το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα ουσιαστικά συζητούμε στο όνομα αυτών που σιωπούν, επειδή ντρέπονται. 1,7 ε, ναι, ε, εκατομμύρια γυναίκες ε, υπήρξαν θύματα βίας πέρυσι, αλλά το 80% δεν καταγγέλουν. Είναι απαράδεκτα φαινόμενα αυτά. Πρέπει να, να λάβουμε νομοθετική δράση η οποία, και να προωθήσουμε νομοθεσία ομοιόμορφη σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αρκούν τα λόγια. Ο προπολογισμό για την καταπολέμηση της βίας είναι χίλιες φορές πιο κάτω από τις ανάγκες. Πρέπει να βάλουμε τέλος ε, ε, στη σιωπή. Αντί να ντρέπονται τα θύματα, θα έπρεπε να ντρέπονται οι θύτες αλλά και η Κομισιόν που μέχρι τώρα δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ελπίζω να αλλάξετε εσείς την κατάσταση κυρία Επίτροπε. Χέντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω στην Επίτροπο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει την Άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει εντό του έτου 2014 μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για την ενίσχυση των ε, εισφορών των κρατών μελών ε, για την καταπολέμηση τη ε, βία σε βάρο των γυναικών και των κοριτσιών που πλήττονται στην Ευρώπη από αυτό το φαινόμενο. Είναι πολύ ενοχλητικό να βλέπουμε να κάθεται με σταυρωμένα χέρια η Κομισιόν. Φυσικά και πρέπει όλα τα κράτη της Ένωσης ε, να επικυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η Κομισιόν πρέπει να, το, ε, να τα πιέσει τα κράτη ε, και θέλουμε το επόμενο έτος να είναι το ευρωπαϊκό έτος της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών ένα πρόβλημα που όλους μας αφορά. Πρέπει να υπάρξει σχετικό πρόγραμμα εργασίας. Και θέλει πλέον η Κομισιόν να μας δείξει πραγματικά ότι βάζει ε, προτεραιότητα ε, το πρόβλημα και την επίλυσή του. Πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει λοιπόν, γιατί ε, εκεί βασίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα το πλαίσιο αυτής της συζήτησης να το αξιοποιήσω για να μιλήσω όχι μόνο για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αλλά και για, τις, ε, για τον, ε, την το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας που αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγική σας παρέμβαση κυρία Επίτροπε πρέπει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε κάθε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Ένωσης το ένταλμα αυτό με το σύστημα της αμοιβαίας αναγνώρισης που είναι εξασφαλιστεί η προστασία από τους παρενοχλούντες εκείνους όταν ε, έρχονται να εγκατασταθούν σε ένα κράτος μέλος. Και επίσης πρέπει από την πρώτη πρώτου του 2015 να υλοποιηθούν αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει σε σχέση με το ένταλμα προστασίας των θυμάτων, γιατί εδώ ακριβώς υστερεί η Ευρώπη ότι αποφασίζει πολλά και ωραία πράγματα αλλά δεν τα υλοποιεί όπως είδαμε και με τι Σύμβαση Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ. Κύριε Καμπεθόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα είναι η διεθνή ημέρα κατά της βίας ε, λόγω φύλου. Και πρέπει να πω ότι στην έναρξη ε, της ε, συνόδου αυτής θα έπρεπε να είχαμε μια επίσημη δήλωση ίσως από τον πρόεδρο ή τέλος πάντων κάποιο θα έπρεπε να είναι εδώ για να μας ευαισθητοποιήσει ε, ένα θύμα γιατί είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Μιλάμε για καταπίεση, καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλοι είμαστε συνένοχοι ίσως και λόγω άγνοιας ή λόγω παθητικότητα αδράνειας. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε αδρανείς ε, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα μπροστά στα φαινόμενα βία κατά των γυναικών. Σε όλη την ιστορία η Ευρώπη, κυρία Επίτροπε, έδειξε το δρόμο προς τα εμπρό για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ε, και δεν πρέπει να αφήσουμε να ε, φύγει η πρόκληση χωρίς να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να προτείνετε παρακαλώ μια σχετική οδηγία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Νόιτσελ, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να απευθυνθώ προσωπικά σε εσά. Πολύ σωστά λέτε ότι και οι άντρες θα πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές της δράσης για να σταματήσει η βία εις βάρος των γυναικών. Ιδιαίτερα, λοιπόν απευθύνω έκκληση σε εσά. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρώτα απ' όλα εσείς προσωπικά πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία στη δράση για να σταματήσει η βία εις βάρος των γυναικών. Εσείς φέρετε την ευθύνη. Εσείς πρέπει να σταματήσετε να κρύβεστε πίσω από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές έχει κληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει επιτέλους μια οδηγία για το πέρας της, βία της βίας της βάρος των γυναικών. Έχουμε να κάνουμε αξιοπρέπεια, με σωματική και ψυχολογική υγεία, με αυτοδιάθεση του σώματος και της γεννητήσιας επιλογής. Εσείς λέτε σήμερα ότι πρέπει να γίνει νέα επεξεργασία όλων των προτάσεων. Εγώ σας λέω το εξής, ότι ήδη έχει γίνει αυτή η επεξεργασία των δεδομένων και πια έχει έρθει η ώρα για δράση. Όποιος καθυστερεί υπερβολικά είναι και υπέτειος. Δεν πρόκειται για ένα πτέσμα μικρής ε, βαρύτητας. Έχουμε να κάνουμε σοβαρότατα εγκλήματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μακέβαν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, Διεθνούς Ανάπτυξης θέλω να μιλήσω για κάτι που δεν έχουμε συζητήσει πολύ. Είναι το θέμα της βίας ε, λόγω φύλου και η καταπολέμησή του μέσω των εξωτερικών μας πολιτικών. Ας πούμε, ε, σε επίγουσες καταστάσεις, πώς μπορούμε δηλαδή να κάνουμε καλύτερα, να, μάλλον να, να, θέσουμε, να δώσουμε τις δυνατότητες στην αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτό το πρόβλημα που είναι γνωστό. Την περασμένη εβδομάδα συνάντησα ανθρώπους που συνεργάστηκαν με και σε τέτοιε καταστάσει που όλοι λένε ότι πρέπει να πάψει η βία σε επίγουσες καταστάσεις. Όσοι δεν έχετε υπογράψει το σχετικό έγγραφο, παρακαλώ να το υπογράψετε. Ε, Αύριο θα δώσουμε το βραβείο Ζαχαρόφα στον ε, ε, δόκτορα Μουγκέμπε που έχει καταπολεμήσει την βία ε, κατά των γυναικών. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα. Ελπίζω πως αυτό θα αποτελέσει μια μαρτυρία στη συνέχιση του έργου του δόκτορα Μουγκέμπε και του χρόνου να μπορούμε να πούμε ότι κάτι καταφέραμε. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία Μορέτη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ αυτή την ημέρα θέλω να ζητήσω από τη νέα Επίτροπο Γιούροβα μια δέσμευση στο να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα και αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή η κοινωνική μάστιγα που ε, πλήττει γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Γυναίκες που ε, υπόκειται σε βία και παρενόχληση και πολύ συχνά αυτές ε, λαμβάνουν χώρα στο πιο ασφαλή χώρο, στο σπίτι, της οικογένειας. Ε, δυστυχώς τα όσα ισχύουν δεν είναι δεσμευτικά για την ώρα ε, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα το οποίο δυστυχώς ε, αυξάνεται καθημερινά. Η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να αφορά μόνο τα κράτη-μέλη μεμονωμένα. Πρόκειται για ένα δραματικό καθολικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να καλέσει μια έντονη συλλογική ευθύνη, πρώτα ηθική και έπειτα πολιτική, και να δεσμεύσει την Ευρώπη σε πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα ξεκινά από μια πολιτιστική εκπαιδευτική εκστρατεία που θα ενημερώσει τις νέες γενιές και που θα οδηγήσει γρήγορα στην υιοθέτηση μιας νέας ε, οδηγίας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. <laughs> Έχω την ε, αδύνατη αποστολή του Catch Έχω 14 που έχουν ζητήσει χρόνο αγόρευσης. Έχετε... Α, συγγνώμη, έχετε μπλε κάρτα για το τελευταίο μιλήτρια. Δέχεστε μπλε κάρτα. Χωρίς μικρόφωνο. Μ' ακούτε, μάλιστα. Κοιτάξτε, άκουσα με προσοχή τα όσα είπατε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε τι λέγεται. Αλλά η οικογένεια ε, είναι πηγή βίας επίσης και δεν άκουσα τίποτα σε σχέση με τη βία που οφείλεται σε θέματα τιμής. Τα εγκλήματα τιμής είναι μέγα πρόβλημα. Το βλέπουμε στη Σουηδία όλο ένα και περισσότερο. Πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα βίας ε, λόγω της τιμής. Ευχαριστώ. Αν επιθυμείτε να απαντήσετε, παρακαλώ, κυρία Μωρέτη. Εγώ πιστεύω πως αυτό το θέμα δεν, αυτή, δεν έχω την ίδια οπτική. Είναι γνωστό ότι η βία που ασκείται κατά των γυναικών είναι ένα πρόβλημα που είναι, εξακολουθεί να είναι βασικά πολιτιστικό. Ε, διακρίσεις που οφείλονται στο διαφορά του φύλου ε, και που γίνονται εντός της οικογένειας, ε, εντός ε, των σχέσεων ανάμεσα σε δύο συζύγους όπου ε, προφανώς ακόμα η γυναική οχυραφέτηση βαραίνει, αλλά το να ορίσουμε αυτά το, αυτού του είδους τη βία ως βία για λόγους τιμής νομίζω ότι το τραβάτε κάπως μακριά και νομίζω ότι είναι ξεπερασμένο. Ε, σας ευχαριστώ, αλλά τώρα περνάει ο χρόνος. Έξι μόνο ερωτήσεις θα δεχτούμε στο ΚΑΤΣΔΙ. Ε, ο κύριος Σαραμπέλα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πραγματικά λίγα έχουμε κάνει και λίγοι άντρε είμαστε εδώ. <laughs> Παρ' όλα αυτά έχουμε εδώ τη λευκή ταινία, τη λευκή κορδέλα. Το είχαν αποφασίσει στην στον Καναδά 25 χρόνια πριν οι άντρε είχε γίνει ένα τρόπο έγκλημα τότε, όπου ένα ε, άνθρωπο που δεν ήταν στα καλά του είχε δολοφονήσει 14 γυναίκε. Ίσως θα έπρεπε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη χρονιά στη βία κατά των ε, γυναικών. <laughs> Στρέφομαι σε εσά κύριε Επίτροπε, διότι με κάποιου συνάδελφου και την Μπάρμπαρα Ματέρα αλλά και με την κυρία Παρμάνοβα, τότε στην Άλντε, με την κυρία Φιγκερέιντο από την ΚΟΕ, με την κυρία Κορνέλη από του Πρασίνου. Πριν τέσσερα χρόνια είχαμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, μια γραπτή δήλωση και ήταν μια από τις λίγες που είχε ε, συγκεντρώσει 402 υπογραφές. Θα πρότεινα να ξαναθέσουμε επιτάπητο σε αυτό το θέμα. Ε, σίγουρα είναι συμβολική η χειρονομία αυτή. Να έχουμε μια γραπτή δήλωση, δηλαδή ελπίζω να έχει ε, την πλειοψηφία των συναντέλφων, να την προσυπογράψουν περισσότεροι από εμάς. Διακόπτεται. Για να έχουμε, επαναλαμβάνω, αυτό το έτο, ολόκληρο έτος για τη βία τον επόμενη, η κυρία Σούκε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Μακρέγκορ αύριο θα, ο κύριος Μουκοέμπε συγγνώμη, θα πάρει αύριο το βραβείο Ζαχάροφ. Και γιατί του απονέμουμε το βραβείο Ζαχάροφ, του γιατρού αυτού, ε, γιατί φροντίζει τις γυναίκες ε, που έχουν αισθήματα ε, κακοποίησης και η Μαλάλα είναι η δεύτερη. Ε, η Επίτροπος Γιούροβα έχει ε, στο χαρτοφυλάκιό της ε, τα θέματα της ισότητας των δύο φύλων. Και ένα άλλο σημαντικό που βιώσαμε σήμερα ήταν η προσφώνηση του Πάπα, ο οποίος μας μίλησε και μας είπε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Αυτό μου δημιουργεί αισιοδοξία. Κάθε χρόνο, 25 Νοεμβρίου, εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και αλλού, έχουμε την ημέρα μνήμης ε, κατά της βίας των γυναικών. δεν θα πρέπει να παραμείνει αυτό συμβολικό. Πρέπει να επικυρώσουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ευχαριστώ. Επόμενος. Επόμενο ομιλήτρια. Μικρό, please. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Στις χώρες μας, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν υπάρχει βία εις των γυναικών, αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνίες δεν έχουν βρει το δρόμο τους. Στην προηγούμενη επαγγελματική μου δραστηριότητα είχα την ευκαιρία να επικοινωνώ με πολλούς ανθρώπους και να συζητώ διαφορετικά ζητήματα, ιδιαίτερα στο θέμα της ε, γενετήσιας βίας, του ελέγχου, της ασφάλειας. Η απάντηση που έπαιρναν πολλές φορές ως προς την βία ήταν ότι ήταν μια παράδοση. Παράδοση που νομιμοποιεί τη βία. Αυτό δεν μπορεί να στέκει όμως σήμερα, δεν μπορεί να στέκει στον 21ο αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αρχίσει να δρά ως κράτος δικαίου και να ενισχύει τις κοινωνίες μας. Δεν έχουμε να κάνουμε νομοθετική δουλειά, έχουμε να κάνουμε με κύρωση της σύμβαση της Κωνσταντινούπολη. Έχουμε να κάνουμε με προγράμματα δράσης. Συζητούμε ένα θέμα που έχει μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να έχουμε μια ε, πολιτική ε, συμφωνία και μεταξύ ε, των πολιτών για να πάψει η βία κατά των γυναικών. Βέβαια δεν βλέπουμε και μια πολύ καλή εικόνα εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί είμαστε πολύ λίγοι όσοι είμαστε εδώ. Πάντω, ε, αυτά τα οποία συζητούμε δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πατριαρχικό φαινόμενο η βία αυτή κατά των γυναικών. Είναι και ιδεολογική και προφορική ε, και ε, κάπως έχει εδραιωθεί μέσα σε, ένα αυτό, μέσα σε ένα σύστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα ε, σε αυτή τη βία να υπάρχει και είναι ένας τρόπος σίγουρα για να διατηρεί τους σχετισμούς δυνάμεων μεταξύ ανδρών και γυναικών γι' αυτό θα ήθελα να εστιάσω στην ανάγκη να υπάρξει κοινωνικός μετασχηματισμός ε, με βάση την ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής και αυτό είναι κατεπήγον. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κλούν για ένα λεπτό. Um, Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το έτος, το Ευρωπαϊκό Έτος για τη Βέκα των Γυναικών είναι ε, μια πρόταση που καλωσορίζω όπως και τη στρατηγική σας ε, για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που λέτε να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την ε, βία λογοφύλου. Είναι σημαντικό όλοι εδώ μιλήσαμε για τη βία κατά των γυναικών, για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο. Πού μπορούμε μεταξύ άλλων να σημειώσουμε πρόοδο. Με την ε, επικύρωση όλων ε, ε, της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλες τις χώρες. Είπατε 8 την έχουν επικυρώσει. Η δική μου χώρα δεν την έχει ακόμη επικυρώσει. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη μου είπε του χρόνου τέτοια εποχή θα το κάνει, γιατί είχαμε προβλήματα με τα σταματικά και τα, μάλλον τα, τα πνευματικά δικαιώματα στο πλαίσιο του συντάγματος. Αλλά αυτό το θέμα είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να μας ε, ανησυχήσει. Οχτώ μόνο χώρες έχουν υπογράψει, έχουν επικυρώσει αυτή τη σύμβαση και είκοσι όχι. Δεν θα ήταν καλό όλε να υπογράψουν, να επικυρώσουν αυτή την σύμβαση. Αυτό θα ήταν ένα καλό βήμα για την καταπολέμηση τη βία ε, κατά τον γενικό σε όλου του τόμου. Τσενίτσκι είναι τελευταία ομιλήτρια. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν υπήρχε χρόνο να δώσω σε άλλου συναδέλφου το λόγο στο πλαίσιο τη διαδικασία αυτή. Signor Σας ευχαριστώ. Η σημερινή συζήτηση δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται ε, στην ημέρα, τη Διεθνή ημέρα της ε, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Είναι ακόμα πολύ σημαντική στη διαστάσεις του φαινομένου σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Στην Ιταλία, στην ετήσια έκθεση για την ε, αυτοκτονία με τα προμελέτης που δημοσιεύθηκε από τη σωτική μας Υπηρεσία την περασμένη εβδομάδα, αποκαλύφθηκε ότι το 2013 σκοτώθηκαν 179 γυναίκες, δηλαδή ένα θύμα κάθε δύο μέρες και σε σχέση με το 12 είχαμε αύξηση της τάξης του 14%. 4% ε, σε τέτοια σοβαρά ε, σε, σε δολοφονίες. Δυστυχώς ε, έτσι είναι και τα στοιχεία, παρόμοια είναι τα στοιχεία στα άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεπής δράση στο, στην προστασία αλλά και στη στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας και των, γυναικών, και των παιδιών των γυναικών αυτών που πολύ συχνά είναι θύματα στη βία αυτή που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ψυχική τους ανάπτυξη. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να υιοθετήσει επιπλέον νομοθετικά μέτρα πέρα από αυτά που ήδη ισχύουν αλλά που προφανώς δεν αρκούν και να ζητήσει την, κύρωση, την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τα κράτη-μέλη και από την ίδια την Ένωση. Σας ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο ώστε να κλείσει τη συζήτηση στην Επίτροπο Γιούροβα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύτιμη και σημαντική συζήτηση που με εμπνέει και μου δίνει δύναμη για τα όσα θα κάνω στην Κομισιόν. Ζητάτε μια νέα πορεία, μια νέα οδηγία. Εγώ έχω την εμπειρία ότι αν επισκεφθώ τώρα εδώ μια νέα οδηγία, θα είναι μια καλή ευκαιρία για να πούμε όλοι, ας περιμένουμε αυτή τη νέα οδηγία. Δεν θέλω να περιμένω, γιατί είναι πλέον ε, ο καιρός για δράση και έχουμε άλλα μέσα εντωμεταξύ πριν να αποφασίσουμε να υιοθετήσουμε μια οδηγία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και φυσικά θα πιέσω για την επικύρωση της, ε, ε, για την κύρωση μάλλον της σύμβάση της Κωνσταντινούπολης καθώς και για ένα πρόγραμμα δράσης, για πραγματική δράση όπου θα υπάρχουν υπάρχει μια ε, στεναρή ανάλυση για τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για το χρονικό πλαίσιο, τη χρηματοδότηση του προγράμματος και τις ε, ευθύνες ε, ε, την ανάθεση ευθυνών. Μην ανησυχείτε λοιπόν, αυτό θα γίνει μέσα στον χρόνο. Μία μόνιμη επίσης εκστρατεία γιατί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μιλήσαμε για τις διάφορες ε, προκλητικές, ε, προκλητικές διαφημίσεις που καταχρώνται την εικόνα της γυναίκας που οι διαφημίσεις σχηματίζουν την κοινή γνώμη. Μπορεί δηλαδή να πει κανείς ότι είναι φυσικό φυσιολογικό να, γίνεται, να, να, να, γίνεται, ε, να ασκείται βία στις γυναίκες ή να γίνεται παρενόχληση. Δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα είναι κάπως προσωπικά αυτά που θα πω. Είπαμε ότι μία γυναίκα κάθε τρεις ε, είναι θύμα βίας. Εγώ θα σας ομολογήσω ότι πριν από πολλά χρόνια υπήρξα θύμα βίας. Και Πολλές φορές στη ζωή μου υπήρξα θύμα προφορικής ε, παρενόχλησης. Δεν θέλω να κάνετε βέβαια τώρα όλοι το ίδιο εδώ, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε ότι εμείς οι ίδιοι που είμαστε τώρα στα ύπαταξιώματα έχουμε περάσει από αυτή την κατάσταση, έχουμε υπάρξει θύματα. Ε, τέτοιων καταστάσεων. Όλα αυτά συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια και θυμάμαι όμως τι αισθανόμουν. Ε, ήταν σαν να ήταν κάπως φυσιολογικό και εγώ ντρεπόμουν για αυτό που μου είχε συμβεί. Αλλά κανονικά πρέπει να ντρέπονται αυτοί οι οποίοι ε, ασκούν βία, όχι τα θύματα τα ίδια. Sorry, last sentence. Before we... Νομίζω λοιπόν ότι πριν ζητάμε μόνο από τους άντρες να αλλάξουν στάση, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τις ίδιες τις γυναίκες, ώστε να μην αισθάνονται, να μην νιώθουν ότι είναι φυσιολογική αυτή η κατάσταση ε, και Προστατέψτε τον εαυτό σας, βοηθήστε μας ε, στις προσπάθειές μας. Ε, με αυτά θα σταματήσω και πραγματικά προσβλέπω στην συνεργασία μαζί σας γιατί πρόκειται για πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ Επίτροπε για τη μεγάλη σας ανθρωπιά και για το ότι είστε τόσο ανοιχτοί όσον αφορά τη δική σας προσωπική εμπειρία βίας. Γιατί όταν ακούμε στατιστικές πρέπει κάποια στιγμή να τα προσωποποιήσουμε όλα αυτά. Είναι δύσκολο βέβαια για σας είμαι βέβαιη, αλλά το εκτιμάμε πολύ. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τέλος της συζήτησης τώρα, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για τις συμβολές σας και το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ε, σφαιρική προσέγγιση της Ένωσης στην μετανάστευση. Έχει υποβληθεί από την Επιτροπή ε, Ελευθερία.